και εφόσον καταθέσει τη σχετική δήλωση ε, συμφερόντων θα αναλάβει θέση στις σχετικές αρχές του Κοινοβουλίου, σχετικά όργανα του Κοινοβουλίου και θα ήθελα επίσης να ακολουθούσε την κυρία